Κύριε Μπέγκε, ε, δύο πράγματα με ενδιαφέρουν. Ε, γραμμή προπολογισμού για το Frontex, για, το, ε, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το άσυλο. Έχουμε βεβαίως ξεχωριστές γραμμές, όμως έχουμε νέες προκλήσεις πλέον. Αντιστοιχούν πλέον αυτές οι γραμμές στις νέες προκλήσεις ή τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τον κύριο Μπέγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πράγματι ε, έχουμε να κάνουμε με, μια ιδιαίτερα, με ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και δύσκολο ερώτημα. Και εφόσον κάνετε αυτό το ερώτημα, επιτρέψτε μου να πω κι εγώ κάτι που ξεπερνάει και την απλή μου αρμοδιότητα του εισηγητή της Επιτροπής μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξής. Στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 14 έως 20, από ό,τι θυμάμαι και εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο, βρίσκομαι από το 89, είχαμε να κάνουμε με τις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις για πολιτές σε δημοσιονομικό πλαίσιο που υπήρξαν ποτέ. Και όλοι μας γνωρίζουμε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο σε πάρα πολλές κατηγορίες ε, είναι στα όρια του και σε τελική ανάλυση το Κοινοβούλιο πλειοψηφικά βέβαια και εξαναγκαζόμενο το Κοινοβούλιο συμφώνησε με το συμβιβασμό διότι στο ανώτατο επίπεδο ικανοποίησαν το δικό μας το έτοιμο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ανάμεσα στα διάφορα δημοσιονομικά έτη. Παράλληλα, στις διαπραγματεύσεις για τον ε, προϋπολογισμό του 2015 είδαμε ότι το ένα επίπεδο, το Συμβούλιο, δεν θυμάται τι ακριβώς έχει συμφωνήσει το άλλο επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ίδια θέματα. Και πρέπει να σας πω σε πάρα πολλά θέματα η Κομισιόν δεν επέδειξε ιδιαίτερο πνεύμα αλληλεγγύης και βοήθειας. Μετά λοιπόν από πολλές ε, διαπραγματεύσεις νομίζω με αρκετά μεγάλη επιτυχία μπορέσαμε να επιτύχουμε διόρθωση του δημοσιονομικού πακέτου προσαρμόζοντας αυτό στο πακέτο Juncker. Βεβαίως εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες αλλά κατορθώσαμε κάποια προγράμματα που έχουν προστιθέμενη αξία όπως ε, τα ε, θέματα των ε, υποδομών, κυρίως μεταφορές και το πρόγραμμα Horizon αυτά να παραμείνουν και να μην εξαφανιστούν. Σήμερα όμως, κατά τη δική μου άποψη, βρισκόμαστε σε κάτι το οποίο ξεπερνάει τις ε, δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα τις ε, δυνατότητες που διαθέτει εδώ και 25 χρόνια. Το τι θα γίνει με τη Frontex και το τι θα γίνει με το Ταμείο για τους πρόσφυγες, ό,τι και να γίνει δεν επαρκεί. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου να μπω στο διατάφτα οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και βεβαίως αν θέλετε μπορούμε να συζητάμε ποιο ώρες, ποιος έφτεξε που. Αυτή όμως η συζήτηση δεν βοηθάει Βεβαίως και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει όταν θα ξεκινήσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάλυση και αξιολόγηση. Δηλαδή όταν ε, θα συζητήσουμε για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, αν θεωρούμε ότι υπάρχει καν τέτοια. Θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον ε, λειτουργούμε σωστά στην αναπτυξιακή μας πολιτική ή μήπως μακροπρόθεσμα θα έπρεπε στην τελευταία να υπάρχουν ε, άλλες πολιτικές για να μην οξύνουμε το δίλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλές από τις γειτονικές μας χώρες και από τις ε, χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Δεν μπορώ να σας δώσω μία ολοκληρωμένη επάρτηση. Ξέρω ότι αυτό απασχολεί πάρα πολλούς ε, συναδέλφους. Εμένα με απασχολεί και κάτι άλλο πάρα πολύ και νομίζω ότι το 2016 πέρα από τις γραμμές του προπολογισμού που θα πρέπει να συζητήσουμε, θα πρέπει να μπούμε στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα έτη. Γιατί ξέρετε, πλέον υπάρχει μια νέα μορφή μετακίνησης λαών, κάτι που κανείς δεν το περίμενε. Έτσι λοιπόν, λόγω των γεγονότων που έχουν προκύψει, τίθεται το εξής ερώτημα. Από κοινού θα διατηρήσουμε τις αξίες μας όπως αυτές ορίζονται στις συνθήκες. Θα παραμείνουμε προσιλωμένοι σε ένα βασικό ερώτημα που αφορά στο δικαίωμα αίτησης θα δεχόμαστε πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες και η τρίτη ερώτηση είναι τι ακριβώς τελικά θα γίνει με μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και τι θα γίνει με προβλήματα που αντιμετωπίζουν τρίτες χώρες που λένε ότι ξέρετε κι εσείς Αγαπητοί, μην δεχτείτε όλους αυτούς γιατί και εμείς θα διάσουμε, δεν θα έχουμε πλέον πολίτες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα δίλημα, τίθεται επιτάπητος η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κατά πόσον δηλαδή θα στηρίξουμε το αξιακό μας σύστημα, κατά πόσον θα παραμείνουμε προσπλωμένοι στις αρχές ε, του ανθρωπισμού ή θα ενδώσουμε σε εκδηλώσεις και εκφάνσεις εθνικιστικού λαϊκισμού. Ξέρετε, όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει με κάποια αύξηση κάποιων γραμμών. Εδώ τίθεται το ερώτημα γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δεν κατορθώσουμε να δώσουμε ικανοποιητικές απαντήσεις, ε, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίω και υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά η Ευρώπη κατ' ουσίαν αποτελείται και συντίθεται από συμβασμούς. Όλοι το ξέρουν. Οι συμβασμοί είναι πόδινοι. Μερικές φορές αναγκάζεται κανείς να δώσει περισσότερα από όσα λαμβάνει. Αν όμως στα ερωτήματα αυτά, όλα αυτά, καταλήγουμε σε φτωχές και πενιχρές απαντήσεις και συμβασμούς, τότε ε, απλώς θα ε, απαντήσουμε στο πώς ε, θα διαχειριζόμαστε το ευρώ, αλλά δεν θα απαντήσουμε στο κατά πόσον παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας. Επ' αυτού πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει τις τελευταίες δεκαετίες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις ε, τροπολογίες ε, της ε, Επιτροπής Προπολογισμών. Αυτές θα τεθούν την Πέμπτη. Καταληκτική μερία και ώρα είναι νομίζω η δωδεκάτη. Λοιπόν, δημοσιονομική πολιτική είναι πολιτική που εκφράζεται μέσα από αριθμούς. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις ε, τρέχουσες ε, προκλήσεις, πώς θα τις ε, συμπεριλάβουμε και μεταφράσουμε σε συγκεκριμένους αριθμούς. Γιατί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και αυτός είναι πάρα πολύ αξιόλογος, αλλά αν θέλετε αυτή είναι μια προαιρετική πρωτοβουλία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη βοήθεια των κρατών μελών. Σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αλλά δεν αρκεί. Γι' αυτό λοιπόν η δική μου παράκληση είναι να προχωρήσουμε πέρα από αυτά που θα ψηφίσουμε σήμερα, να διεισδύσουμε στην ουσία της ύπαρξης και της δυνατότητας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απολύτως απαραίτητο αυτό γιατί οι εξελίξεις σε πάρα πολλά κράτη-μέλη με καθιστούν ιδιαίτερα ανήσυχο γιατί αν το τρένο συνεχίσει με αυτό το ρυθμό φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα διάλυσης και καταστροφής όλων αυτών που επιτύχαμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Διαδικαστικό. Αλλά δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Δέκα λεπτά πριν την ψηφοφορία και πολύ ευθραδός τα είπε ο συνάδελφος. Ε, θα ήθελα να ζητήσω 90 δευτερόλεπτα για να απαντήσω ε, σε αυτά. Όχι σήμερα, μια άλλη μέρα πριν από την επόμενη ψηφοφορία. 90 δευτερόλεπτα να έχω στη διάθεσή μου. 15% δηλαδή του χρόνου που δώσατε στο συνάδελφο. Εγώ ήρθα για να ψηφίσω εδώ πέρα. Δεν ήξερα ότι θα έχουμε δεκάλεπτες ομιλίες ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Α, να το κάνω τώρα. Ωραία. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα επιλύονται καλύτερα και προσδιορίζονται πολύ καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα είναι η πλήρης αδυναμία και η ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει οτιδήποτε που να έχει κάποια σημασία. Η μετανάστευση είναι πολύ επίμαχο ζήτημα, αλλά να κάνω ένα σχόλιο για τη χώρα μου. Ένα σχόλιο απλά. Με βάση στατιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσίας πριν από τρεις ημέρες στη χώρα μου που είναι λιγότερο από τη μισή ομοσπονδιακή δημοκρατία. Έχουμε δεχθεί 8 εκατομμύρια μετανάστες από το 1997 και μετά, όταν η κυβέρνηση των εργατικών έκανε ένα πολύ επικίνδυνο πραγματικά ε, πείραμα που δεν είχε τη συμφωνή γνώμη των Βρετανών. Μέχρι 4 εκατομμύρια Σύρους μετανάστες, πρόσφυγες πρέπει να δεχθεί και άλλους από την Αφρική. Θα μπορούσαμε να τα δούμε ε, με μεγαλύτερη ε, νυφαλαιότητα όλα αυτά, αν δεν είχαμε λάβει ήδη 8 εκατομμύρια. Σχεδόν ολόκληρο το πληθυσμό της Ιδίας ή της Δανίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συνένεση. Συνένεση δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει συνένεση, γιατί έχουμε παταγώδη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν σε όλους τους ε, τομείς. Ξεκινάμε με το ευρώ, που είναι ε, η καταδίκη της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, που προκαλεί μόνο Και ακούμε τώρα 10 λεπτά μία ομιλία που ουσιαστικά συνιστά πλήρη άρνηση της πραγματικότητας. Είχατε τα 90 δευτερόλεπτά σα, ε, κύριε συνάδελφε. Δεν έχουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή, λέει ο πρόεδρο. Και υπερβαίνουν οι συζητήσει που είχαμε και τι αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα. Δεν είναι σίγουρα καθόλου άστοχη αυτή η συζήτηση. Δεν πρέπει να γίνει όμω τώρα. Α περάσουμε στην ψήφιση τη νομοδότηση ε, για τον προπολογισμό του 2016. Ξέρετε ότι θα ψηφίσουμε καταρχάς τις τροπολογίες ε, της γνωμοδότης και μετά θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες του σχεδίου έκθεσης, του σχεδίου προβλήματος για το 2016. Δύο έχουμε λοιπόν, δύο λίστες ε, ψηφοφοριών. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης αρχικά. Τροπολογία 5. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, σαφές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τροπολογία 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ψήφι πέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 4, περνάμε στην τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2 που καλύπτει τις τροπολογίες 4 και 6, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογία 8, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 8. Αν ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίας, η τροπολογία 8 απορρίπτεται. Επόμενη, η τροπολογία 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 12. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 12. Πάμε στην τροπολογία 11. Καταπίπτει 11. Πού πηγαίνουμε. 13, 4, 16, right? 13. 13 4, 16. Uh, next is amendment number 16. 16. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά εποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά προτιμώ να ελέγξουμε τη συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 23, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο Τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Θα γίνει ηλεκτρονικά ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή και τώρα προχωρούμε στη δεύτερη λίστα ψηφοφορίας. Δημοσιονομικές τροπολογίες, τροπολογίες από του προπολογισμού. Πρώτη είναι η τροπολογία 6600, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Έχουμε τώρα μια προφορική τροπολογία και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από το καλοκαίρι συζητήσαμε για το θέμα αυτό και τότε, στο τέλος της συζήτησης, είχαμε πει ότι λόγω της πολιτικής μας ανάλυσης επιθυμούμε να υπάρξει αύξηση αυτών των κονδυλίων. Παράλληλα όμως ε, δεν ήταν ε, σωστή αυτή η σχέση ε, που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές και είχαμε πει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αποθεματικό. Τώρα όμως το αποσύρω αυτό το αποθεματικό γιατί εντωμεταξύ η Κομισιόν μας έπεισε, μας έδωσε αρκετά επιχειρήματα για το ότι είχε κάποια προβλήματα με κάποιους εταίρους. Τώρα μας είπε ότι λύθηκαν αυτά τα προβλήματα. Άρα δηλαδή στην συμβαστική πρόταση 4 εξετάσαμε το θέμα αυτό και γι' αυτό προτείνω τώρα να αυξηθούν τα κονδύλια όπως προβλέπετε αλλά να μην δημιουργήσουμε απαραίτητα αποθεματικό. θα του αποθεματικού. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δεν ξέρω, συμφωνείτε όλοι με αυτή την προφορική τροπολογία. Πολύ ωραία. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για την προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενο είναι η 6601, καταπίπτει αυτή η γραμμή. Πάμε στην 62-6602. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, Προτιμώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την 6602. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Τώρα, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και εγκρίθηκαν οι τροπολογίες στη γνωμοδότησή μας. Ευχαριστούμε τους αδέλφους, ευχαριστούμε τον εισηγητή και έτσι ολοκληρώνεται σήμερα η ηλεκτρονική ψηφοφορία για σήμερα. I will take a moment uh, to wait for the... Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Thank you.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 Can we resume our meeting, please? So, thank you very much. Uh, Να συνεχίσουμε παρακαλώ τη συνεδρίασή μα. Σα ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο για το σημείο 7 της μέση διάταξη. το ρόλο δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση εντό των για την καλύτερη επίτευξη των στόχων εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνάδελφο Σκά Κέλλερ που έχει συντάξει την γνωμοδότηση από του Πρασίνους. Θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση. που αφορά την διάσταση επενδύσεων και εμπορίου εντός του συστήματος των Εθνών και όπως είπα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας την κυρία Σκά Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πράγματι είχα την ε, ευχαριστήση να συντάξω αυτή τη σύντομη γνωμοδότηση. Γνωρίζετε ότι οι γνωμοδοτήσει είναι περιορισμένε ό,τι αφορά την έκτασή του, είναι άρα ε, σύντομοι, αλλά μπορείτε να κάνετε στο δυνατόν περισσότερα σχόλια. Ο κύριος Πάβο Βέρινεν είναι ο αρμόδιος για την Καθήλυνη Επιτροπή, αρμόδια Επιτροπή, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μιλάμε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των ΗΠΑ, ίσως να μην σα έρχεται ε, σε αυτό το πλαίσιο το εμπόριο αμέσως στο μυαλό. Είναι σημαντική πτυχή όμως, είναι σημαντικό σκέλος ε, και απασχολεί τις επιτροπές, ε, τις ομάδες εργασίας και τα ψηφίσματα των Εθνών. Είπε ο κύριος Μπέγκε επίσης ότι έχει να κάνει και με τις αναπτυξιακές πολιτικές. Το εμπόριο λοιπόν είναι σημαντικό στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής στο πλαίσιο των Ηνωμένων και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έτος 2015 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά του στόχου της ανάπτυξης ε, που θα θετηθούν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχουμε επίσης τη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα στο Παρίσι αργότερα φέτος και όλα αυτά έχουν μεγάλη σχέση και με το εμπόριο. Πράγματι, το εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά αν ε, τα πράγματα δεν πάνε καλά, μπορεί να είναι και αρνητικός ο ρόλος του εμπορίου. Πρέπει να δούμε και τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Μεγάλες οι ε, για το εμπόριο αυξάνει δυνητικά τέλο πάντων μπορεί να αυξήσει τι εκπομπέ με τον τον άλλο τρόπο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση στην εμπορική μα πολιτική. Το εμπόριο μπορεί επίση να επηρεάσει και προκλήσει όπως είναι η πιστιστική κρίση που είχαμε το 2008 με πολλά εκατομμύρια ε, ανθρώπους στον πλανήτη να πεινάνε. Και η δυσλειτουργία των αγορών ή ο ρόλος των αγορών ήταν κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η εμπορική πολιτική της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι να την παρακολεί. Αυτό είναι το πνεύμα που διέπει τις προτάσεις μας, τις συστάσεις μας στο πλαίσιο αυτής της γνωμοδότησης. Να αναφέρω ορισμένε από αυτές τις συστάσεις ε, αφορά μία από αυτές την φοροποφύγη και φοροδιαφύγη. Έχουμε την ε, έκθεση UMSATS για την ανάπτυξη πριν από το ε, καλοκαίρι δημοσιεύτηκε και μας έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη ε, τάση για φοροδιαφυγή και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, να γίνουν ε, οι δέουσες μεταρρυθμίσεις, επίσης φύλλο και εμπόριο. Έχουμε ένα πρόγραμμα ε, στο, στο πλαίσιο των ΗΠΑ για μέτρα που θα δεν αφήνουν στο περιθώριο τις γυναίκες αλλάζει η οικονομία, αλλάζουν και οι ρόλοι και θα πρέπει να υπάρξει πραγματική ισορροπία μεταξύ των φύλων και η πολιτική θα πρέπει και αυτή να ασχοληθεί πιο ενεργά με την εφαρμογή μέτρων ε, για τον τομέα αυτό. Θα πρέπει να είναι ε, ένα κριτήριο και βέβαια ξέρετε ότι δεν μπορούσα να πω πιο πολλά γι' αυτό και να αναφέρω μια τρίτη σύσταση. Επτά είναι τον αριθμό επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη ο ΙΕ έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είναι στη διαδικασία της ε, ε, περαιτέρω συγκεκριμενοποίησης ε, αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. Και θα έπρεπε αυτές να είναι δεσμευτικές για τις εμπορικές συμφωνίες ιδίως ε, της Ευρωπαϊκής και ένας μεγάλος ε, πρωταγωνιστής ε, και εταίρος μας είναι και οι ΗΠΑ που έχουν πολλές συμφωνίες εμπορικές με διάφορες χώρες. Έχουμε λοιπόν και την έκθεση Επιτροπής ΑΦΕΤ που μιλά για ένα συμβούλιο βιώσιμης ανάπτυξης όπως το ΙΕ. Μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον εισηγητή. Και το θέμα της συνέπειας και συνεκτικότητας μεταξύ εμπορίου και πολιτικής ανάπτυξης και αναπτυξιακών στόχων. Θα ήθελα να παρακαλώ στους αδέλφους να διαβάσουν την γνωμοδότηση και να την εμπλουτίσουν με τις ιδέες τους και τις τροπολογίες τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου αλλά και τη γραμματεία που με βοήθησε σημαντικά για την κατάθεση αυτής της, ε, αυτού του σχέδιου γνωμοδότηση πριν το καλοκαίρι ώστε να την έχετε ήδη αναχείραση. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε. Και τώρα καταρχήν οι σκιώδεις εισηγητές. Από το ΕΛΚ ε, έχουμε τον Τζιν Κέλλη, ε, ε, τον κύριο Μάουλορ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σύντομο το κείμενο όμως υπενθυμίζει σημαντικά πράγματα όπως το πόσο προσιλωμένοι είμαστε ε, στο πολυμερέ σύστημα και το σύστημα του ΟΗΕ. Γι' αυτό θα χαιρετήσω και το ερώτηση της συναδέλφου Κέλλερ. Επίσης, ε, πολύ θετικά ε, αντιμετωπίζουμε τις συστάσεις να ληφθούν υπόψη και οι πολιτικοί στόχοι του ΟΗΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ μέρος της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών χαίρομαι που δεν ξεχάσατε δύο προτάσεις ε, που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα σώμα. Την καταπολέμηση της φοροποφής και φοροδιαφύγης αφενός, που είναι στο επίκεντρο σήμερα ε, του ενδιαφέροντός μας και θα χρειαστεί να νομοθετήσουμε ή τέλο να γνωμοδοτήσουμε γι' αυτό το ζήτημα στους επόμενους μήνες και επειδή υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ μας για αυτό το θέμα, χαίρομαι που αναφέρεται και το, τη μόνιμη επιτροπή ή μόνιμο δικαστήριο που αν βέβαια ε, συγκροτηθεί θα ενταχθεί στο σύστημα του ΟΗΕ και θα πρέπει να σέβεται τις αρχές του πολιτικού συστήματος και αυτό είναι πολύ ε, καλό. Να επιστήσω όμως την προσοχή σας σε δύο πρόσθετα σημεία. Το πρώτο είναι ότι θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε την η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσωτερικά και εξωτερικά με την εμπορική της πολιτική θα πρέπει να δεσμευτεί υπέρ της ε, ε, εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και το δεύτερο σημείο είναι οι εμπορικέ συμφωνίε που υπογράφουμε με τρίτε χώρε, ιδίω στι λιγότερο αναπτυγμένε, θα πρέπει να είναι δίκαιε και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των χωρών αυτών με βάση ε, του ε, αναπτυξιακού στόχου τη χιλιετία. Αυτά είναι τα στοιχεία και ίσως ε, θα καταθέσουμε από την ομάδα μας ε, τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πάρα τη συντομία του, να επαναλάβω το κείμενο, είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για τη δουλειά της κυρίως ε, γιατί έπρεπε να την επεξεργαστεί την έκθεση κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και αυτό σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Νομίζω είναι σημαντικό ως Επιτροπή Διεθνού Συμπορίου να τοποθετηθούμε σε αυτήν την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων παρότι αισθάνομαι ότι ε, ο ρόλος που τους έχει αποδοθεί είναι λιγάκι υπερβολικός κυρίως όσον αφορά το ε, διεθνές ε, δικαστήριο, κάτι που προτείναμε πριν από το καλοκαίρι στο πλαίσιο του ψηφίσματος TTIP. Βεβαίως έπρεπε να ληφθεί μια τελική απόφαση. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης αξιολόγηση πριν τελικά αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Επιπλέον δεν νομίζω ότι γίνεται επαρκής αναφορά στη σημασία και το ρόλο των επενδύσεων για την ε, ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια. Νομίζω αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη πρόσβαση σε, σε επενδύσεις και εμπόριο, να χρησιμοποιήσουμε όλους τους υπάρχοντες μηχανισμούς, έτσι ώστε αυτές οι χώρες επιτέλους να αποκτήσουν τις επενδύσεις που χρειάζονται απελπισμένα. Εν πάση περιπτώσει αισθάνομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο να γίνουν περισσότερες επενδύσεις κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτά να ισχύσουν και όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δραστηριοποιηθεί και δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία χρόνια και αυτό οδήγησε σε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των επενδύσεων. Να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τις αγορές έτσι ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την παγίδα της φτώχειας να τις βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν δύσκολες συζητήσεις και με εμά τους ίδιους για τη γεωργία, για τις επιδοτήσεις, για το πώς θα συνεχίσουμε ή θα σταματήσουμε σε αυτούς τους τομείς, αλλά πιστεύω στη δύναμη του εμπορίου για να ε, μην υπάρχει πια φτώχεια και για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να επανέλθουν ε, στον ε, στη δραστηριοποίηση που χρειάζονται. Εγώ λοιπόν προσβλέπω στην κατάθεση τροπολογιών, θα καταθέσω τροπολογίες και ελπίζω να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, μέσα από το εμπόριο, όπως σας είπα. Και εμεί ευχαριστούμε η Μαρίκε Σάκε εκ μέρους των φιλελευθέρων. Θα το δω στις λεπτομέρειές του το κείμενο αργότερα. Το έχουμε συζητήσει με την ΑΦΕΤ. Νομίζω ότι επειδή είμαι και μέλος της ΑΦΕΤ θα το κοιτάξω και εκεί το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει σημαντικότερο ρόλο ε, στο πλαίσιο ε, των Ηνωμένων Εθνών, τη δουλειά της Κακέλερ ε, θα τη δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα επανέλθω το συντομότερο δυνατόν. Εκ μέρου ε, της, EFTD, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξή. Την κυρία Σκέλετ τη θεωρώ μία από τα καλύτερα μέλη αυτή τη επιτροπή. Αυτό πρέπει να το πω. Είναι μεγάλη τιμή για μας να την έχουμε μέλους. Αλλά φοβάμαι ότι δεν συμφωνώ με αυτά που μας λέει. Θέλω βέβαια πρώτα απ' όλα να πω σε τι συμφωνώ. Και ε, συμφωνώ κυρίως σε αντίθεση με τον εκπρόσωπο της CCR στο θέμα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να προβληθεί αυτός ο μηχανισμός. Επίσης ε, συμφωνώ με το να υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη ε, να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Πολύ καλύτερα αυτό από πρωτοβουλίες που θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Η δική μου χώρα έχει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και παρότι αυτή η έδρα απειλείται συνεχώς, εμείς την έχουμε αυτή την ε, θέση και έχουμε και δικαίωμα βέτο. Εδώ έχουμε 28 επιτρόπους και δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα βέτο. Είναι λοιπόν λυπηρό ε, το ότι ο εκπρόσωπος της CCR που είναι και εκπρόσωπος ε, του κυβερνώντος κόμματος στην πατρίδα μου μοιάζει να μην τα εκτιμά όλα αυτά αλλά έχουν οι καιροί γυρίσματα. Μπας περιπτώσει, να πω κάτι για την εμπορική πολιτική. Πολύ σωστά ελέγχθη και το έγραψα αυτό που ελέγχθη για να μην το διαστρεβλώσω. Ε, είπε ο εκπρόσωπος της ECR ότι το εμπόριο είναι ένας τρόπος για να αναπτυχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, είπε η εκπρόσωπος της ECR. Το θέμα είναι ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να καλύπτει τα πάντα. Η εμπορική πολιτική είναι απλά ένας τρόπος για να πει κανείς ότι εγώ έχω πολύ ιδιαίτερους στόχους και θέλω να χρησιμοποιήσω το εμπόριο ως εργαλείο, για, ως όπλο για να τους ε, επιτύχω. Εντάξει, αλλά πρέπει κανείς να ξέρει περί τίνος πρόκειται και το θέμα είναι ότι αν αποδίδει κανείς ε, στο εμπόριο όλη αυτή την ε, τεράστια σημασία των στόχων του, τότε παρεμποδίζεται το εμπόριο και έχουμε λιγότερο εμπόριο. Αυτό επηρεάζει τους αναπτυσσόμενους. Δεν λέω να συμφωνήσετε μαζί μου, απλά θέλω να πω ότι γίνεται πλέον μεγαλύτερη πολιτικοποίηση του εμπορίου. Αυτό έχει επιπτώσεις και κόστος και απλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και τέλος ε, θέλω να πω και το εξής. Δεν θα επανέλθω στα επιχειρήματα για το TTIP δεν θα τα ξαναπούμε πάλι όλα αυτά που έχουν υποθεί, αλλά θέλω να πω ότι κατά τη δική μας άποψη υπάρχει ένας τομέας όπου συμφωνώ στο σημείο 5 που λέτε ότι το Διεθνές Δικαστήριο θα πρέπει να είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Καλύτερα εκεί λοιπόν από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν τελείως διαφορετική νομοθεσία από αυτή που έχουμε στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως ε, υπάρχει μια καινούργια πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την εκπροσωπώ εδώ σήμερα. Ε, ε δυστυχώς από τις συνθήκες Λισαβόνα και μετά, το 2009 και μετά, έχουμε ε, μία εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για εξωτερικά θέματα και πολύ φοβούμαι ότι η δράση που έχει αναλάβει έκδοτη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιτίθεται ουσιαστικά στους δεδηλωμένους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η φτώχεια και η καταπολέμησή της ε, στις νότιες χώρες ναι να τις βοηθήσουμε αλλά για να τις βοηθήσουμε θα πρέπει επιτόπου να προσφέρουμε τη βοήθειά μας πλήττει σήμερα η κρίση την Ευρώπη. Έχουμε την απειλή της Διατλαντικής Συμφωνίας και με όλα αυτά τα δεδομένα φοβόμαστε ότι θα έχουμε αξιμένες ε, ε, δυσκολίες στη γυρία Ήπειρο των 28 ε, χωρών. Θα πρέπει χωρίς να κάνουμε κοινωνικό ντάμπινγκ ούτε και φορολογικό να βοηθήσουμε επιτόπου αυτές τις χώρες. Είδαμε δυστυχώς τι συνέβη με το Πακιστάν, με το εργοστάσιο που κάηκε. Είχαμε βάσει συμφωνιών αναγκαστεί να ε, θυσιάσουμε ένα κομμάτι της κλωστοϊφαντουργίας ε, στην Ευρώπη. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν μπορούμε μέσω αυτής της εξωτερικής πολιτικής να έχουμε και νέες αγορές για τις γαλλικές παραδείγματος χάρη επιχειρήσεις, αλλά προσοχή, δεν μπορούμε να θυσιάζουμε ε, στο βωμό της εξωτερικής πολιτικής τις επιχειρήσεις και την οικονομία της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε. Ζητώ συγγνώμη από την αλλά δεν είχα ε, κανένα σκιώδη εδώ στον κατάλογο μου, γι' αυτό ε, χάλασα τη σειρά με την οποία ε, συνήθως δίνουμε ε, το λόγο. Λέει ο κύριος Σόλς, δεν πειράζει πρόεδρε, έτσι έχω την ευκαιρία να παρέμβω μετά το συνάδελφο από τη νέα πολιτική αυτή ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφος Κακέλερ για τη δουλειά που έχει κάνει και θέλω να τονίσω πως για πρώτη φορά, από τότε που εγώ είμαι εδώ τουλάχιστον, που η ΙΝΤΑ έχει τη δυνατότητα να αποφανθεί για την ετήσια έκθεση ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς τον ΟΗΕ. Σχόλιο εκτό μικροφόνου. Συνεχίζει ο κύριο Σόλτ. Ναι, πρώτη φορά γίνεται η συλλογή νομοδοτήσεων από όλε τι επιτροπέ για να εμπλουτιστεί αυτή η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεύτερον, ευχαριστώ την εισηγήτρια, διότι προσπαθεί να ε, επικεντρωθεί ε, στα πιο ουσιαστικά ζητήματα. Δεν είναι αυτονόητο αυτό στην ε, ΑΦΚΟ Προσπαθούμε κάθε φορά όταν ε, εκδίδουμε μια γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι καθήλυνα αρμόδια να επικεντρωνόμαστε κι εμεί στα βασικότερα ζητήματα. Στην Επιτροπή ΙΕΝΤΑ επίση θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ρόλο τη εμπορική πολιτική ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζοντα ότι υπάρχει αυτό το σύστημα στον ΟΗΕ ισόρροπη εκπροσώπηση των κρατών αλλά και των περιφερειακών οργανώσεων. Ως περιφερειακή οργανώση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιπρόσθετα δικαιώματα. Βάσει της χάρτας του ΙΕΠ έχουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε κι εμείς, ε, ούτως ώστε μέσω του ΟΗΕ να συμβάλλουμε στην ε, ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Λοιπόν, ας πάρουμε ε, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, την υφαρπαγή γης ε, στην Αφρική, παραδείγματος χάρη και τις μη επιδοτούμενες ε, γεωργικές ε, καλλιέργειες ε, και τη διατήρηση των εθνικών αγορών θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε μέσω της εμπορικής μας πολιτικής υποστηρίζοντας τα τοπικά προϊόντα των τρίτων αυτών χωρών και όχι αντικαθιστώντας τα με τα δικά μας. Ελπίζουμε ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή δεν θα καταψηφίσει τις γνωμοδοτήσεις άλλων επιτροπών όπως έγινε δηλαδή με την TTIP. Θα προσπαθήσει να ενσωματώσει λοιπόν ελπίζουμε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη σοφία των ε, υπόλοιπων επιτροπών και έτσι ελπίζουμε να συμβάλλουμε σε αυτήν την εξαιρετική έκθεση που συντάσσει η Εξωτερικών Υποθέσεων για το σύστημα ε, λειτουργίας του ΟΗΕ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα περνούμε στα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ροντρίκε Πινιέρο. Έχει... Θα πάρετε εσεί το λόγο. Ναι, όχι, γι' αυτό απευθυνόταν στου μεταφραστέ. Ευχαριστώ. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση της. Πράγματι, εστιάζει στο διεθνέ εμπόριο και σίγουρα ε, δεν είναι, όπως είπε και η ίδια, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για τον ΟΗΕ. Αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη έκθεση γιατί δεν μπορεί η ανθρώπινη ανάπτυξη να εννοηθεί χωρίς ε, το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο που θα εργάζεται όμως για την ε, βελτίωση, την ανάπτυξη των ανθρώπων. Δεν μπορεί να είναι αυτό σκοπό το εμπόριο. Και θα πρέπει να δούμε και υπό ποιε συνθήκες παράγονται και τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τη δυστυχία που δεσπόζει τον κόσμο δυστυχώς. Θα ήθελα τώρα να τονίσω τρεις πτυχές που αναφέρονται στην έκθεση και που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σχολιάσω, να αναπτύξω περαιτέρω. Πρώτον, Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες από τον ΟΗΕ και από όλα τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για την καταπολέμηση των παραβίασεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τροφοδοτούνται από συγκεκριμένε εμπορικέ πρακτικέ. Δεν πρέπει να λησμονούμε ένα ζήτημα που απασχόλησε την Επιτροπή μα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή ε, τις, ε, την εξόριξη μεταλλευμάτων από εμπόλεμες περιοχές, από περιοχές που βρίσκονται σε εμπόλεμη ζώνη ή από πρακτικές επιχειρήσεων που καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εμπόριο όπλων βέβαια και άλλα. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και την προαγωγή της στρατηγικής για την ε, αξιοπρεπή εργασία που προωθεί η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και νομίζω ότι και στον ΟΗΕ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η φωνή μας και ως ένας και ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακούγεται πέρα αυτή τη στρατηγική και τη πρόθεση τη. Δεύτερον, κάτι εξίσου σημαντικό, ο ρόλο των επιχειρήσεων και η εταιρική, κοινωνική εταιρική ευθύνη. Πρέπει να φέρετε ρητά, θα ήθελα τουλάχιστον, ε, ο ρόλο που πρέπει να διδραματίζουν σε αυτόν τον τομέα όλε οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου, κατά πολέμηση τη φοροδιαφυγή και καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Ο ΙΕ έχει το ρόλο του, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τη σειρά τους πρέπει να το κάνουν γιατί υπάρχουν φορολογικές, φορολογική παράδειση, γιατί ε, τους, τους στηρίζουν και κάποιες κυβερνήσεις. Τέλος, η ισότητα των φύλων. Δράτω με τις ευκαιρίες για να πω ότι λυπούμε βαθύτατα όπως ψήφισαν οι πολιτικές ομάδες της δεξιάς, ως αποτέλεσμα να καταψηφιστεί μια δική μας τροπολογία, με την οποία ζητούσαμε να γίνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να δούμε τι αντίκτυπο έχει η διάσταση του φίλου, συμπερίληψη τη διάσταση του φίλου στο έθνες εμπόριο. Αυτά είχα να πω ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι τώρα στα μέλη της Επιτροπής μας. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να διατυπώσει κάποιο σχόλιο, αν όχι να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον βέβαια κρίνει ότι πρέπει να σχολιάσει κάτι. Αν όχι θα ακολουθούμε την ε, ΣΚΑ, ε, την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Όντως μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Πρέπει να περιοριστούμε στι δικέ μα ορμοδιότητε όμω, γιατί υποβάλλουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Δίκαιη τη έκθεση, αλλά όντω. υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορούμε να συμπεριλάβουμε και μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ε, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις ε, για τους στόχους ε, του εξωτερικού εμπορίου. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. 3 ε, μέχρι τι 6 το απόγευμα. Αυτή είναι η προθεσμία για την υποβολή ε, τροπολογιών και στις 21-22 Σεπτεμβρίου θα γίνει συζήτηση για την έγκριση της έκθεσης. Θα ήθελα και να σας ενημερώσω για να, έχετε, δει να το ξέρετε κι εσείς, λοιπόν, 21-22 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνουμε το τελευταίο σημείο, το σημείο 7 στη Μέση Διάταξη και τώρα περνούμε στο τελευταίο σημείο ανθρώπινα δικαιώματα στη διαπραγματεύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Ε, είναι ένα αίτημα προφορικής απάντησης για τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ε, διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Στην αρχή της συνεδρίασής μας ε, αναφέρθηκα στην ε, ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα αυτό το μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επί της αρχής έχουν καταλήξει συμφωνία με το Βιετνάμ για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Είναι εξαιρετικά αυτά τα νέα. Επίσης, θα θυμάστε ότι είχαμε μεταβεί τον Απρίλιο ε, ένα, ένα μεγάλο κλιμάκι της ε, Επιτροπής μας πήγε τον Απρίλιο στο Βιετνάμ για να συζητήσει τις διαπραγματεύσεις και τη μελλοντική συμφωνία. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το ζήτημα. Θα δώσω το λόγο στην συντάκτρια αυτής της προφορικής ερώτησης, ε, η κυρία Σάλκη από τους φιλελεύθερους. Πρόεδρε, να σας πω ότι χαίρομαι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Βιετνάμ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι διαπραγματεύσεις πλέον ολοκληρώθηκαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και επίκαιρη η προφορική ερώτηση. Ένα από τα ερωτήματα που θέτουν πολλοί άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών αλλά γενικότερα από το ίδιο το Βιετνάμ είναι ακριβώς αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Η εμπειρία του παρελθόντος ε, σε σχέση με τις εμπορικές ε, συμφωνίες ε, δείχνει ότι μπορεί σαφώς να βελτιωθεί η ευμάρεια των πολιτών ε, το εμπόριο είναι ένα από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, πρέπει όμως να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ε, τις ανησυχίες που υπάρχουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτή λοιπόν η προφορική ερώτηση αναζητά το πώς μπορεί να πληροφορηθεί καλύτερα για το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει και έλεγχος μετά την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και όλα αυτά για να μην επιτρέψουμε στο να επισκιαστεί αυτό το τόσο σημαντικό θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την επιτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Πολύ ωραία λέει ο συνάδελφος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ΕΛΚ, οι σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, ε, εκτιμάμε ιδιαίτερα τη δουλειά αυτή που έχει γίνει για την ε, σύναψη εμπορική συμφωνίας με το Βιετνάμ. Θέλω όμως να πω το εξής. Όσον υπάρχει το θέμα σύναψης μιας εμπορικής συμφωνίας, αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να επισημάνει κανείς και το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με ορισμένα θέματα που για μας είναι σημαντικά. Ε, σε αυτά λοιπόν ε, που υπόθηκαν από τους ε, συναντέλφους θέλω να προσθέσω ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τώρα που έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία τι θα γίνει τελικά όχι μόνο με τα αμυγός οικονομικά θέματα αλλά τι θα γίνει και σε σχέση με τη δυνατότητα βελτίωσης που θέλουμε να υπάρχει σύντομα βελτίωση λοιπόν όσον αφορά γενικότερα την κατάσταση των πολιτών αλλά και μια σειρά αξιών που για μας ε, είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες. Πρέπει να υπάρχει το ελάχιστο επίπεδο δικαιωμάτων για τους πολίτες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα, κυρίως για τη χώρα που συζητάμε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και να δοκιμάσουμε οτιδήποτε υπάρχει έτσι ώστε να ενισχύσουμε τον έλεγχο και ο έλεγχος να είναι σαφέστερος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρους τώρα της ΓΚΟΕ Λοιπόν, χίλια συγγνώμη, δεν είδα. Στην ECR θα δώσω το λόγο, στην Emma Clarke. Προσωπώ τη συνάδελφο λοιπόν είναι και μόνος εισηγητή για το Βιετνάμ, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Ως μόνιμος εισηγητής λέει λοιπόν ότι χαίρομαι πολύ που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής ε, μετά από δυόμιση χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων ε, την πρώτη του είδους ε, που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αναπτυσσόμενη χώρα και δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του εμπορίου για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δημιουργία πλούτου από τι δύο πλευρέ και θα βελτιώσει σχέση των οικονομιών και θα δημιουργήσει νέε δυνατότητε πρόσβαση σε υπηρεσίε και επενδύσει. Ό,τι αφορά τώρα την προφορική ερώτηση τη συναδέλφου Σάκε, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ε, ουσιαστικά ε, προβλέπει ότι θα πρέπει και τα ανθρώπινα δικαιώματα δημοκρατία, το κράτος δικαίου να συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα θέμα που πρέπει να παραμείνουν στη σχεδιάταξη μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι την τελική έγκριση. σύμφωνα ότι θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση, βοήθεια, να χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι δεν αφορά το άρθρο 3 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρισιμότητα των εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει να είμαστε πιο ε, προσεκτικοί, διότι οι σχέσει μεταξύ απελευθέρωση εμπορίου και σεβασμού των δικαιωμάτων είναι πολύπλοκοι δεν είναι εμπόδιο στο εμπόριο η αιρεσιμότητα. Πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβαδίζουν αυτά τα δύο, εμπόριο δηλαδή και σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το εμπόριο πρέπει όμω να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, να μειώνει τη φτώχεια, γιατί η φτώχεια, η καταπολέμηση τη φτώχεια είναι ε, σημαντική για την πράσινη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεύτερον, πρέπει να εφαρμόσει τη αρχή τη διαφάνεια, να υπάρχουν δεσμεύσει, στόχοι στο πλαίσιο των συμφωνιών ε, ελεύθερου εμπορίου για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιμένουμε και συγκεκριμένε απαντήσει από την Κομισιόν. Uh, και τώρα από την ΚΟΕ. Ε, εκπροσωπώ την Ελεονόρα Φρέντσε που δεν, μπορεί να έρθει, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, δυστυχώς. Υποστηρίζουμε αυτή την προφορική ερώτηση και ε, μας εξέπληξε αυτό που μάθαμε από, μάθαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι επί της αρχής ε, ε, ε, έχουν καταλήξει συμφωνία για μια έχουν επί της αρχής καταλήξει συμφωνία για την σύναψη αυτής της συμφωνίας σε ελευθερό εμπόριο. Πρώτα απ' όλα διότι έχουμε τις ε, αντίθετες συστάσεις από τον ΟΗΕ και βάσει των πληροφοριών που έχουμε δεν έχουν συμπεριληφθεί τα πετούμενα χέρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αυτό το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη που δεν έχει κανένα ε, ουσιαστικό αντίκτυπο, αλλά αυτό δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο θα συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, τα συμβαλόμενα μέρη ο... και έχουμε, έχουν απαγγελθεί κριτικέ κατά του Βιετνάμ για διάφορα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την ισότητα των δύο φίλων για να φέρω μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ε, από τις ειδικέ διαδικασίες του ΕΕ αλλά και από την διαμεσολαβήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε στοιχεία βάσει των οποίων υπάρχει παραβίαση σαφέστατη των ε, του άρθρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ολομελία δεν έχει γίνει ανοιχτή συζήτηση σε σχέση με τους εφιστάμενους μηχανισμούς για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της, ε, των συμφωνιών ελευθερού εμπορίου. Ε, πέρα από τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν και τα εργατικά δικαιώματα. Υπάρχει το σχετικό κεφάλαιο στη Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τι απαιτήσει, όμω ε, δεν βλέπουμε ε, καμία προστασία σε σχέση με την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων μέσα στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε του οδηγού όχι μόνο σε αυτά τα ηχέγγυα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για τα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα, διότι εκεί εντοπίζεται ένα σοβαρό αντίκτυπο των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Χρειάζεται λοιπόν παρακολούθηση και αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθηση τη συμμόρφωση με τι υποχρεώσει για αυτά τα δικαιώματα. Τώρα ε, για του ε, πράσινου θα ακούσουμε τη Σκά Κέλλερ. Σα ευχαριστούμε, ε, ευχαριστούμε του φιλελευθέρου για αυτή την ερώτηση που υποβάλλανε. Όντω είναι επίκαιρο το ζήτημα και συμφωνούμε με τον προσανατολισμό που ακολουθείτε για την αιρεσιμότητα θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και το μόνο που θα θέλαμε να προσθέσουμε είναι επίσης, όπως ακούσαμε τώρα, η εξολόγηση αντικτύπου για την κατάσταση ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας ελευθέρω Εμποδίευη. Το 2014 το ζήτησε το Κοινοβούλιο μέσα σε ένα ψήφισμα ότι η εξολόγηση αντικτύπου για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται και η διαμεσολαβήτρια επίσης ε, ε, ζήτησε αξιολόγηση αντικτύπου. Πολύ δύσκολα μπορούμε να δούμε πώς το άρθρο 21 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει σεβαστό εάν λείπει αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό θέλουμε να συμπεριληφθεί στη συμφωνία. Οι εμπειρογνώμονε του ΟΗΕ έκαναν μελέτε και εξέτασαν ακριβώ αυτό το ζήτημα, πώ το εμπόριο και οι επενδύσει. Αυτές μάλλον οι συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων επηρεάζουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς μπορεί να γίνει η αντίστοιχη αξιολόγηση και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις θέσεις όταν συντάσσει ε, την εμπορική της πολιτική. Επίσης, ε, αναφέρθηκαν και τα πολιτικά συμπεράσματα, πώς μπορώ εγώ να καλωσορίσω και να επικροτήσω αυτά τα πολιτικά συμπεράσματα, αν δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό του. θα μπορούσε ίσω μας, να μα ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουμε αρνητική εμπειρία εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι μα λέτε Α, όχι, είναι τεχνικά αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό τα ρυθμίζουμε, αλλά τελικά έχουν ε, ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτήρα. Μόνο έτσι μπορεί να εμπλακεί ενεργά το Κοινοβούλιο στη διαδικασία. Εάν λοιπόν έχει καταλήξει σε συμφωνία από τις αρχές, ε, το κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο τελικό κείμενο. Το τμήμα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη επίσης ε, ε συγγνώμη για την ε, ε, συμφωνή κράτους επενδυτή ε, δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στην ε, συμφωνία. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για αυτό το ζήτημα, αλλά εν γέννη αυτό το θέμα των πολιτικών συστάσεων δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και θα θέλουμε να ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Η FTT, η ΕΝΕΠ, δεν έχουμε κανέναν. Έχουμε όμως ε, δύο συναδέλφους, Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε την συνάδελφα Λυσία, θα ασχοληθώ και εγώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό συνδέεται εξάλλου με την προηγούμενη συζήτηση για τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα για την ετήσια έκθεση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώ ενισχύονται αυτά μέσα από την εξωτερική πολιτική. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Βιετνάμ και συστηματικά θα θέτουμε αυτό το ζήτημα ε, για ε, τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου δεν μπορούμε να θυσιάζουμε ανθρώπινες ζωές. Ε, στο Ράνα Πλάτσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει κατάφορες παρεμβίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πέρα από το ζήτημα της αιρεσιμότητας θα πρέπει να θέσουμε ένα σοβαρότερο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταγγελία και παρακολούθηση περιπτώσεων παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε εργαλεία ε, διαλόγου και συνεργασίας ναι μεν, αλλά αυτά δεν είναι ε, δεσμευτικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να στραφούμε προς σταθερούς μηχανισμούς υποβολής ε, καταγγελιών και παρακολούθησης αυτών των καταγγελιών με δεσμευτικά αποτελέσματα. Έχουμε δαπανίσει πολλή ενέργεια σε σχέση με το κεφάλαιο για τις επενδύσεις ε, σε αυτές τις συμφωνίες. Αν αντίστοιχα ασχολούμαστε και με το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσως θα είχαμε κάτι έτσι πιο ρηξικέλεπτο αλλά και αποτελεσματικό. Σας ευχαριστούμε. Η Τζούτ και τον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Κοιτάξτε, Νομίζω ότι αν δεν αναφέραμε με απόλυτη σαφήνεια τη θέση του διαμεσολαβητή για το Βιετνάμ, αυτό θα ήταν λάθος. Γιατί ο διαμεσολαβητής ε, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λειτουργήσε κακόπιστα. Και αν θέλετε αυτό είναι μια δρυμύτατη κριτική έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στο κείμενο της προφορικής ερώτησης γιατί αλλιώς αν δεν το κάνω αυτό θα ήταν μεγάλη παράληψη. Ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να ασκήσει μεγαλύτερη ε, πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν επιτιμεί κανείς άλλο το λόγο. Ε, στρέφομαι λοιπόν τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την Χέλενα Κιούνιχ, την ε, Διευθύντρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ξεκινώντας θέλω να πω, ε, επιβεβαιώνω και επαναλαμβάνω αυτά που έχουμε πει και κατά παρελθόν, ότι είναι πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην εμπορική πολιτική και κυρίως είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε όλες τις κοινοτικές πολιτικές για να ενισχύσουμε τη σημασία και της εμπορικής πολιτικής. Και αυτό να το κάνουμε με ένα συνεπή τρόπο να χρησιμοποιούμε όλες τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και μεγάλο καιρό και πολύ καιρό είναι καθοριστικής ε, σημασίας ε, και όσον αφορά τις συζητήσεις για εμπορικά θέματα. Γενικότερα βέβαια για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εμπορική πολιτική. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος, πολλές εκδηλώσεις και με πολλές ευκαιρίες είναι καλύτερα να υπάρχει μια πολιτική συμμετοχής αντί για μια πολιτική που εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο σε προαπαιτούμενα. Και όσον αφορά την FTA, εμείς πρέπει να σας πω, ε, θεωρούμε ότι εδώ έχουμε ένα πολύ ισχυρό κεφάλαιο και σε αυτό το κεφάλαιο το οποίο καλύπτει διάφορα εργατικά θέματα αλλά και άλλα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Υπάρχει και μία σχέση ανάμεσα στην FDA και τις απαραίτητες ρήτρε τη Συμφωνία Συνεργασίας την οποία έχουμε ήδη συνομολογήσει με το Βιετνάμ. Επιπρόσθετα λοιπόν ε, σε αυτό το συσχετισμό έχουμε και μία συγκεκριμένη υποδομή ε, για το, την αηφόρο ανάπτυξη που σημαίνει ε, τη συνεργασία των αρμόδιων επιτροπών και από τις δύο πλευρές οποτεδήποτε προκύπτουν σχετικά θέματα και βεβαίως τα πρακτικά αυτών των επιτροπών θα διετίθενται αμελητή. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη συναντήση αυτών των επιτροπών. Όσον αφορά τώρα την ουσία του θέματος, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να απαντήσει οποτεδήποτε το θέμα έρθει στην Ολομέλη. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά την FDA, ε, θα έχετε διαπιστώσει ότι έχουμε ήδη εκδώσει ένα σημείο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Σας έχουμε δώσει ε, και σε εσά λεπτομέρειες. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να εξετάζουμε ε, κάποια ε, στοιχεία που έχουν σχέση με την νομιμότητα και τον ομότυπο των κειμένων. Θα σας στείλουμε τα κείμενα το συντομότερο δυνατόν όταν θα έχουν λάβει τελική μορφή όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αξιολόγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι έχουν γίνει ήδη αρκετές συζητήσεις και όπως ξέρετε, ένας από τους ε, λόγους που δεν αποφασίσαμε να, κάνουμε, να προβούμε σε ειδική αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό είναι μια ευρύτερη πολιτική. Η αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2012 έγινε σε όλα τα κεφάλαια, πάντα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτή η αξιολόγηση με το Βιετνάμ έχει ήδη γίνει. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν θα επαναλάβει μία τέτοια αξιολόγηση. Έχω σίγαση. Έχω σίγαση. Δες το. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του διαμεσολαβητή, θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή ε, Βεβαίως, ε, αν θέλετε ευχαρίστως να δημοσιεύσουμε τι περιλαμβάνει αυτή η επιστολή του διαμεσολαβητή. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα επανέλθω τώρα στην εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους να που έλαβαν Σίγουρα δεν απαντώνται με αυτή την προφορική ερώτηση όλα τα αναπομένοντα ερωτήματα και δεν καλύπτει όλες τις συζητήσεις που θα πρέπει να έχουμε για τις διαπραγματεύσεις αυτές και τις μελικές συμφωνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μελετήσαντε ε, τη συμφωνία όταν έρθει η ώρα. Σίγουρα δεν μπορούν να λυθούν όλα τα κακά στο Βιετνάμ με όρους, υπερπροθέσεις ή με σχετικές ε, αναφορές στο διεθνές εμπόριο. Βλέπω όμως ότι συμφωνεί δεξιά και αριστερά ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και δεν είναι και σύνθεση φαινόμενο αυτή η συνένεση στην Επιτροπή μας. Να σας δώσω τώρα ορισμένες λεπτομέρειες για την διαδικασία. Πρώτον, πρέπει να επικαιροποιηθεί το προτινόμενο κείμενο με βάση ε, τις ε, πραγματικότητες αυτής της ε, συμφωνίας επί της αρχής και επί οι πολιτικές ομάδες θα μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες ή ήδη κάποιοι ανέφεραν ε, Τη ε, τροπολογία του Ζητώ όμως να γίνει και μια τεχνική συνάντηση, αφού έχουμε αυτές τις τροπολογίες, για να ε, καταρτήσουμε την προφορική ερώτηση και σίγουρα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το ευρύ φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ορισμένοι εστιάσατε συγκεκριμένα στι συνθήκες εργασία και άλλα κοινωνικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα σχόλια του ΕΣΥΑΡ για το ανθρώπινο δικαιώματα και το εμπόριο που συμβαδίζουν, συμφωνώ απόλυτα και Νομίζω ότι αυτή η δέσμευση είναι καλή και δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Ελπίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη βάση για να έχουμε ένα κείμενο που ικανοποιεί όλου του συναδέλφου και βέβαια μετά να προχωρήσουμε ε, στο άμεσο μέλλον σε μια συζήτηση με την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. 21-22 Σεπτεμβρίου θα προβλεφθεί συζήτηση του θέματος αυτού. Ε, Επομένω εδώ ολοκληρώνουμε και το σημευτό και έχουμε άλλα δύο ζητήματα. Το εννέα που είναι τα διάφορα. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, εγώ έχω ένα σύντομο θέμα να θέσω υπόψη σας για τους ε, βουλευτές, ε, τους συνεργάτες ε, και την γραμματεία να ευχηθώ να έχουμε πολύ καλές αυθινοπορεινές εργασίες και κυρίως για την επόμενη σύνοδο και να σας πω για το 10 της προσεχής Συνεδρίασης, ότι η επόμενη Συνεδρίαση μας θα είναι 21 Σεπτεμβρίου 3 με 6.30 και 22 Σεπτεμβρίου πρωί και απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνω η συνάντησή μας. Ευχαριστώ.